procederemos a las declaraciones del consejo y de del consejo de asuntos exteriores. στις ε, Συμβουλίου και Κομισιόν για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ε, Εξωτερικών για την ειδική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Η κυρία Μάλμστρομ εκ μέρου του Συμβουλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι. Η σύγκρουση στην ε, Μέση Ανατολή ήταν κάτι το οποίο είχαμε συζητήσει και στην αρχή της Σουηδικής ε, Προεδρίας και επανερχόμαστε τώρα να κάνουμε μια ανασκόπηση. Και ο Καλ Μπίλτ ήταν στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων την προηγούμενη εβδομάδα, ο Υπουργός των Εξωτερικών, πρώην Υπουργός των Εξωτερικών, και την προηγούμενη εβδομάδα το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών υιοθέτησε συμπεράσματα και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για το ότι και τα 27 κράτη-μέλη υποστηρίζουν τα συμπεράσματα που αποσαφηνίζουν τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ειρηνευτική διαδικασία. Με τα συμπεράσματα αυτά, Συμβούλιο και Προεδρία θέλουν να αποστείλουν ένα σαφές και ευρωπαϊκό μήνυμα ε, να πούμε πώς ελπίζουμε πώς θα επαναληφθούν οι συζητήσει μεταξύ των εταίρων στο μέλλον. Ανησυχούμε πράγματι για την έλλειψη Πρόοδο στην ειρηνευτική διαδικασία. Επίσης ξεκαθαρίσαμε πω υποστηρίζουμε τι προσπάθειε των ΗΠΑ για ειρήνευση. Καλούμε εμεί τα μέρη να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για ζητήματα όπως η Ιερουσαλήμ, τα σύνορα, η ασφάλεια κτλ. Συνεχίζουμε λοιπόν τις συζητήσεις που είχαμε επμακρών. Οι θέσεις μας βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και τις έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, είναι σαφής θέση μας, πρέπει να υπάρξουν δύο κράτη με βάση τα σύνορα του 1967 και να είναι οριστική η λύση και για την Ιερουσαλήμ και για τα σύνορα όσον αφορά την Ιερουσαλήμ. Λέμε πως εάν πρόκειται να επιτευχθεί η ειρήνη πρέπει να λυθεί το ζήτημα της Ιερουσαλήμ ως κοινής πρωτεύουσα των δύο κρατών μέσω διαπραγματεύσεων. Η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων Ισραήλ-Παλαιστινίων σχετίζεται και με το ζήτημα των επικισμών. Πρόσφατα είπε πως θα υπάρξει μια μερική πάυση των επικισμών το Ισραήλ. Καλωσορίζουμε αυτή την απόφαση και ελπίζουμε να συνεισφέρει στην επανάληψη διαπραγματεύσεων που θα έχουν νόημα. Σημειώνουμε με κάποια ανησυχία την απόφαση την πρόσφατη απόφαση της ε, κυβέρνησης του Ισραήλ στις 13 Δεκεμβρίου να επαναλάβει την οικοδόμηση οικισμών σε περιοχές εθνικής προτεραιότητας, κάτι το οποίο παντιβαίνει την προηγούμενη της απόφαση και δεν δημιουργεί βεβαίω σωστή απόφαση όταν ο συνάδελφός μου κ. Κάλσον ήρθε εδώ πέρα στην Επιτροπή Ανά... μου κυρία Κάλσον ήρθε εδώ πέρα στην Επιτροπή Ανάπτυξης ε, μίλησε για τις εξελίξεις που υπάρχουν επί τόπου και για τη στήριξη που πρέπει να δοθεί και ειδικά όταν μιλάμε για την Ανατολική Ιερουσαλήμ, για τους επικισμούς, για την πρόσβαση στη Γάζα. Είναι υποσχέσεις αυτές τι οποίες κάναμε και τους τελευταίους μήνες είδαμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Προεδρία ξεκαθάρισαν την θέση μας για το ζήτημα των επικισμών και για την απομόνωση της Γάζας η απομόνωση της Γάζας είναι απαράδεκτη και αντιπαραγωγική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επανέλαβε το αίτημά της να ανοίξουν τα συνοριακά φυλάκια χωρίς όρους για ανθρωπιστική βοήθεια αγαθά και ανθρώπους. Επίσης να εφαρμοστεί το σχετικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να γίνει σεβαστό το ανθρωπιστικό δίκαιο. Επίσης αυτοί οι οποίοι κρατούν τον Γκυλάντ Σαλίτ, τον Ισραηλινό στρατιώτη, πρέπει να τον απελευθερώσουν και κάποια ε, λόγια τώρα για τη Γάζα. Η Αίγυπτος και ο Αραβικός Σύνδεσμος προσπαθούν να αποφύγουν ένα διχασμό μεταξύ Γάζας και Δυτικής Όχθης ε, του Ιορδάνη. Ελπίζουμε να υπάρξουν ελεύθερες εκλογές όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, γιατί ένα είναι σαφές η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί εάν οι Παλαιστίνοι είναι ενωμένοι. Οι διπλωμάτες μας επιτόπου παρακολουθούν την κατάσταση στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και η άποψή τους είναι πως το Ισραήλ ε, προσπαθεί να εξασθενήσει την Παλαιστινιακή παρουσία εκεί πέρα. Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ανατολική Ιερουσαλήμ, να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής των Παλαιστινίων και είναι σαφές το μήνυμα στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Επίσης θα πρέπει να θυμόμαστε πως πρέπει να βρεθεί και μία λύση με την, με την Συρία και με το Λίβανο από πλευράς Ισραήλ για να έχουμε ειρήνη στην περιοχή και υποστηρίζουμε τις πρόσφατες δηλώσεις που έγιναν που θα έχουν πτωση λίγο την περιοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που ζητήσατε να γίνει και αυτή η συζήτηση. Ε, σας ευχαριστούμε κυρία Μάλστρον. με ώρα της Επιτροπής, το λόγο να δώσουμε στην κυρία Άστο. Um, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Συμβούλιο, όπω ελέγχθη, ενέκρινε διάφορα σημαντικά συμπεράσματα για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή την περασμένη εβδομάδα. Καθορίζω στη βασική μα θέση σε μία σειρά από κρίσιμα θέματα και κατά την άποψή μου αυτό έγινε με ένα αποφασιστικό και σαφή τρόπο. Δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία ε, είπε η Πρόεδρο, ε, ούτε τα συμπεράσματα. Πάντω θα ήθελα να σα πω ότι βεβαιώντα τι αρχέ μα, ελπίζω να, μπορέσα, να μπορέσαμε να βοηθήσουμε στην αποκατάσταση τη εμπιστοσύνη ε, των Παλαιστινίων να επιστρέψουν στην ερευνητική διαδικασία. Βεβαίω τα συμπεράσματα αυτά θα βοηθήσουν ιδιαίτερα και εμένα, γιατί με αυτόν τον τρόπο ε, θα έχω μια σταθερή βάση για να προχωρήσω του προσεχεί μήνε. Ε, με καλέσατε για να μιλήσω για την, πολιτική, για την εργασία σε πολιτικό επίπεδο και για την κατάσταση στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Ε, Μα απασχολεί ιδιαίτερα, διότι είναι κατεχόμενη περιοχή μαζί με το υπόλοιπο τη δυτική ε, όχθη. Ε, διαφωνούμε με, το, με, το, με, το, με την κατεδάφιση των σπιτιών των Παλαιστινίων, με, τον, με τη δημιουργία επικισμών και με ε, το τείχος διαχωρισμού. Ε, όλα αυτά τα αναφέρουμε ε, σε πολιτικό επίπεδο, σε διπλωματικό επίπεδο με τις δημόσιές μας δηλώσεις. Ταυτόχρονα όμως προσπαθούμε με πρακτική συνδρομή προς, προς τον Παλαιστινιακό πληθυσμό στην Ανατολική Ιερουσαλήμ να βοηθήσουμε την κατάσταση. Για παράδειγμα, λείπουν 1.200 σχολικές αίθουσες για τα παιδιά των Παλαιστινίων στην περιοχή. Τους βοηθάμε λοιπόν για να βρουν εγκαταστάσει για την εκπαίδευση. Επίσης, σε επίπεδο νοσοκομείων θέλουμε να διατηρηθούν τα νοσοκομεία στην περιοχή αυτή. Επίση, βοήθεια προ του νέου ε, που υποφέρουν από πολύ ψηλά ποσοστά ανεργία και από σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Σήμερα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ 4,6 εκατομμύρια ευρώ ε, ε, δαπανούμε για τι συγκεκριμένε δραστηριότητε. Ένα άλλο θέμα αφορά την κατάσταση στη Γάζα. Επανειλημμένα ε, προσπαθούμε να βοηθήσουμε και ανησυχούμε ιδιαίτερα για τι συνθήκε διαβίωση του Παλαιστινιακού λαού στην περιοχή αυτή. Εδώ και πολύ καιρό οι δωρητέ δεν μπορούν να προβούν σε έργα νοικοδόμηση. Υπάρχουν βασικά προβλήματα, για παράδειγμα έλλειψη καθαρού πόσιμου νερού. Πρέπει να ανοίξει τα περάσματα το Ισραήλ χωρί καθυστέρηση για ε, γιατί πρέπει να αναπτυχθεί ο ιδιωτικό τομέα και να μειωθεί η εξάρτηση από τη βοήθεια τη περιοχή αυτή. Ήρθε η στιγμή τα συμπεράσματα του Συμβουλίου να τα θέσουμε ε, σε πρακτική εφαρμογή. Και πρέπει τώρα να σκεφτούμε το πώ θα ξεκινήσουμε μια νέα πολιτική διαδικασία. Οι δύο πλευρέ αυτή τη στιγμή έχουν απομακρυνθεί περισσότερο όσον αφορά τη δέσμευσή του ε, ε, για την ειρηνευτική διαδικασία. Προσεχώ θα μεταβώ στην περιοχή, θα προσπαθήσω να συναντηθώ και με τι δύο πλευρέ και να δούμε το πώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αποτελέσει το μοχλό τη αλλαγή. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούν με την βασική προτεραιότητα ε, της αποκατάστασης και της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων των δύο πλευρών. Διαπραγματεύσεις όμως ουσιαστικές, όχι προς χάρη των διαπραγματεύσεων. Διαπραγματεύσεις που θα, ορίσουν, που θα, που θα οδηγήσουν σε μια καινούρια σελίδα. Δεν μπορούμε πλέον να ανεχθούμε ένα νέο γύρο άκαρπων διαπραγματεύσεων. Ε, κοιτάξτε, εδώ και πολλά χρόνια ξεκινούν και σταματούν οι διαπραγματεύσει, ξεκινώντα ε, με το Σεπτέμβριο του 1993, ε, όταν υπογράφηκε η βασική αρχή συμφωνία για την αρχή των διαπραγματεύσεων. Αυτά μα πλέον δεν έχουν νόημα. Το θέμα είναι να τεθούν όλα τα ζητήματα επιτάπητο, συμπεριλαμβάνοντα και το καθεστώ τη Ιερουσαλήμ ω μελλοντική κοινή πρωτεύουσα. Και όλα αυτά βεβαίω μέσα σε ένα συμπεφωνημένο χρονικό πλαίσιο. Θέλουμε σοβαρέ δεσμεύσει και πολιτική βούληση και από εκ εκ μέρου του Ισραήλ και εκ μέρου τη Παλαιστίνη, έτσι ώστε να υπάρξουν γνήσιε ε, και πραγματικέ διαπραγματεύσει. Εμεί θα βοηθήσουμε και τι δύο πλευρέ για να αναλάβουν τη δέσμευσή του και θα του υποστηρίξουμε στο δύσκολο δρόμο των διαπραγματεύσεων. Εγώ θα φροντίσω έτσι ώστε ε, οι διαπραγματεύσει αυτέ και οι συνομιλίε να γίνουν με αρμονικό τρόπο. Ε, επανειλημμένα ε, ε, τους έχουμε δώσει την ευκαιρία να διαπραγματευτούν διμερώς. Εμείς το, προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε την Παλαιστινιακή Αρχή για την οικοδόμηση των θεσμών. Άρα λοιπόν μπορούμε να τους βοηθήσουμε, και, και, αλλά σήμερα... Η, Παλαιστίνη είναι διαιρεμένη και σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε πρακτικό επίπεδο. Αξιόπιστε διαπραγματεύσει όμω απαιτούν ένα ισχυρό εταίρο εκ μέρου τη Παλαιστίνη. Ε, το Ισραήλ όμω δεν θα χάσει από ένα ισχυρό εταίρο και συνομιλητή. Ε, το Ισραήλ ε, προέβη σε, ε, ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση παγώνοντας τους επικισμούς. Πάντως εξακολουθεί να παραμένει ο βασικός πρωταγωνιστής για τις διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή. Και να σας πω ότι ήρθε η στιγμή όλα αυτά να γίνουν πραγματικότητα συντονίζοντας τις θέσεις μας ως προς τη στρατηγική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει, να υποστηρίζει τις προσπάθειες αυτές και το κουαρτέτο το οποίο πρέπει πρέπει ε, ε, να το αναβιώσουμε. Ε, το απαιτεί η ανάγκη για ειρηνευτικέ διαπραγματεύσει. Το κουαρτέτο μπορεί να αποτελέσει την σωστή διαμεσολάβηση η οποία απαιτείται. Κοιτάξτε, η Μέση Ανατολή απαιτεί συνολική λύση και εδώ θα παίξει σημαντικό ρόλο και η Συρία και ο Λίβανο. Περιμένουμε με ανυπομονησία την υλοποίηση τη πρωτοβουλία, ειρηνευτική πρωτοβουλία εκ μέρου των Αράβων. Η προσέγγιση μα θα πρέπει να είναι και περιφερειακή αλλά και πολυμερή, έτσι ώστε να συμπληρώνεται το διμερέ επίπεδο επίπεδο συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης. Θα ε, είμαστε σε στενή επαφή ε, του προσεχεί μήνε και ξέρω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να παίξει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο και με την ιδιότητά του ω αρχή του προπολογισμού. Ε, οι αντιπροσωπείε μα εργάζονται στενά με το Νομοθετικό Συμβούλιο των Παλαιστινίων και με την Κνεσέτ. Την ε, ε, περασμένη εβδομάδα ε, μια αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τα κατεχόμενα και ανέφερε τι ανησυχίε τη για την κατάσταση επιτόπου. Τέλο, θα ήθελα να καλωσορίσω τη συνέχιση τη ομάδα εργασία του Κοινοβουλίου για την Ειρηνευτική Διαδικασία και θα ξανασυναντηθούμε αυτή την εβδομάδα. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, και τώρα να περάσουμε στις πολιτικές ομάδες. Εκ, εκ μέρους του ΕΛ και δύο λεπτά το λόγο έχει ο κύριος Κασουλίδης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης νέων Παλαιστινίων ηγετών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγινε μια βαθιά συζήτηση για την ειρηνευτική διαδικασία, μια λύση και τη λύση μία λύση σε δύο φάσεις. Επί τη βάση των συνόρων του 67 με την Ιερουσαλήμ ως ε, πρωτεύουσα αμφωτέρων, αποστρατικοποίηση του Παλαιστινιακού κράτους, επανάληψη της ε, αραβικής συνευτικής πρωτοβουλίας, εγγύησεις ε, έξωθεν και μία αλλαγή του δημογραφικού χαρακτήρα του εβραϊκού κράτους. Ενώ λοιπόν οι νέοι έχουν ένα ενιαίο όρομα, οι ενήλικες ακόμα τσακώνονται. Η Αιγυπτιακή Πρωτοβουλία ε, για την Παλαιστινιακή κατάσταση στο να υπάρχει ένα ακόμα εκρεμή και η κατάσταση στη Γάζα με τους ε, φυλακισμένους Τζιλάτ και Σαρίμ συνεχίζεται. Σύμφωνα με την ε, αναφορά του επικεφαλής ε, της αποστολής του ΟΗΕ η κατάσταση στη δική ε, Γερουσαλήμ γίνεται, ε, στη Όχθη γίνεται όλο και πιο δυσάρεστη. Από την άλλη, το Ισραήλ, μια δημοκρατική χώρα, δίνει λίγη σημασία στις βλάβες που προκαλεί στα μάτια της διεθνούς κοινότητας και περιορίζεται μόνο σε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κασουλίδη. Κύριε κυρία Άτκινς έχει το λόγο. Κύριε Άτκινς, ζητήσατε το λόγο ε, στα πλαίσια του Catch the Eye ή ε, ε, για να κάνετε μια ερώτηση προς τον κύριο Κασουλίδη. Catch the Eye, μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα το λόγο έχει εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και των Δημοκρατικών για δυόμιση λεπτά ο κύριος Βόμποτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε του Συμβουλίου, κυρία Αντιπρόεδρε της Κομισιόν. Να σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για την πρωτοβουλία σας. Ήταν θετική πρωτοβουλία και σας συγχαίρω και ευχαριστώ την κυρία Άστον για το ότι στην πρώτη συμφάνιση εδώ πέρα κάθεται στην πλευρά της Κομισιόν Οπότε, ε, εντάξει, όταν μιλάμε για εξωτερική πολιτική, όσο να μην έχει τόση σημασία που κάθεστε, σημασία έχει να έχουμε μια κοινή εξωτερική πολιτική. Δεύτερον, η δήλωση του Συμβουλίου νομίζω πως είναι θετική συμβουλή και δεν είναι καθόλου αντι-Ισραηλινή. Κάθε άλλο είναι προς το συμφέρον του Ισραήλ, της ασφάλειας, του Ισραήλ, της σταθερότητας, του Ισραήλ. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Γιατί εάν εμείς ως Ευρωπαίοι δραστηριοποιούμαστε, πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια αυτή της δραστηριότητα. Θέλω να σα παρακαλέσω κυρία Άστον πραγματικά να το προσέξετε αυτό. Τις επόμενες... Ε, κάποιες μέρες συζητήσαμε πριν από λίγες μέρες με συναδέλφους ε, με, από το Κογκρέσο τον ΗΠΑ όπου δεν υπάρχει καμία αντίληψη για το τι συμβαίνει με τους Παλαιστίνιους. Αντιλαμβάνονται τις θέσεις του Ισραήλ πλήρως, θέλουν να σταματήσει η τρομοκρατία, να πάει ο στρατιώτης πίσω στην οικογένειά του, αλλά εξακολουθούμε να εμείς να αντιλαμβανόμαστε και την άθλια κατάσταση των Παλαιστινίων ειδικά δε όσον αφορά τα σύνορα του 67, ειδικά όσον αφορά την δύσκολη κατάσταση στην Ιερουσαλήμ, ειδικά όσον αφορά την κατάσταση με τους επικισμούς. Βλέπουμε πως υπάρχει εδώ πέρα μία διπλή στάση. Μία λένε σταματάνε, μία συνεχίζουν. Μετά πάει στο πρόγραμμα εθνικών προτεραιοτήτων. Μετά μιλάνε για την φυσική εξέλιξη και συνεχίζουν να επεκτείνονται. Κόβουν στα δύο Παλαιστινιακούς οικισμούς και συνεχώς τους παίρνουν γη. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο. Αυτό το οποίο συνέβη και με την ε, κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία, νομίζω πως, θα το πει και ο συνάδελφος ο κύριος Ντερόσα, νομίζω έχουμε δικαίωμα ως βουλευτές να πάμε στη Γάζα και να δούμε τι γίνεται. Τι έχει να κρύψει το Ισραήλ να μην το δουν οι βουλευτές στη Γάζα. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε από κοινού τον αγώνα. Νομίζω η διαφάνεια είναι ε, βασικό ζήτημα εδώ πέρα και πρέπει να το υποστηρίξουμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε, Ευχαριστώ, κύριε Σμπόβοδα. Εξ ονόματος των Δημοκρατών και Φιλελευθέρων για δυόμιση λεπτά το λόγο έχει η κυρία Νίτς Ιτεμπρεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε είπατε εκπρόσωπε, με συγχωρείτε. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου. Θα ξεκινήσω με εσά, ε, κύριε. Μάλλον θέλω να συγχαρώ στο πρόσωπό σα ολόκληρη την Σουηδική Προεδρία για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και γενικότερα και ειδικά για την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Ελπίζω πως είναι σημαντικό μήνυμα για τις μελλοντικές εξελίξεις για όσους βλέπουν πως για πρώτη φορά η έκθεση των επικεφαλής ε, των αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορώ πλέον να το πω αυτό, εφόσον έχουν περάσει συνθήκη της ε, Λισαβόνας, έχουν εγκριθεί από όλους. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο. Δεύτερον, πως και τα συμπεράσματα που παρουσιάζονται, ε, παρουσιάστηκαν από την Σουηδική Προεδρία έγιναν δεκτά σε σχέση με την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Είναι λοιπόν ένα σημάδι αυτό για τις μελλοντικέ εξελίξεις και ελπίζω πως θα αντιληφθούν πόσο σημαντικό είναι αυτό οι Ισραηλινές αρχές, πόσο σημαντική είναι αυτή η εξέλιξη. Γιατί, συνάδελφοι, εμείς συζητάμε για τη Μέση Ανατολή εδώ και τόσους μήνες και καμιά φορά μοιάζει πραγματικά με συσήφια αυτή η υπόθεση, ένα βήμα μπρο και δύο προς τα... στα πίσω κάνουμε. Υπάρχουν ε, λόγια ελπίδα αλλά και πολύ περισσότεροι λόγια απελπισία. Οπότε και για την ομάδα μου είναι αυτονόητο πως και το Ισραήλ και η Παλαιστίνη θα πρέπει να μπορέσουν να ζήσουν γειτονικά σε δύο χωριστά κράτη με ειρήνη και θα είναι εγγυημένη ασφάλεια και των ε, δύο. Και για πρώτη φορά συμφωνούμε όλοι σε αυτό και συμφωνούμε ποια είναι τα βήματα τα οποία θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Η Ιερουσαλήμ είναι μία από τις ωραιότερες πόλεις του κόσμου και πάνω από την Ιερουσαλήμ, το φως της Ιερουσαλήμ είναι κάτι το εκπληκτικό. Είναι απίστευτα τραγικό όμως ο κόσμος ο οποίος μένει εκεί δεν μπορεί να το χαρεί γιατί φοβάται να βγει και να χαρεί αυτό το φως και ελπίζω λοιπόν τις μέρες αυτές των Χριστουγέννων να τα καταφέρουμε να δώσουμε μια όψη στην ειρήνη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Ιτεμπρόκ. Εξ ονόματος των Πρασίνων και της ε, ε Ελεύθερης ε, ε, Ευρωπαϊκής Συμμαχίας η κυρία Λούκας έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θέλω να καλωσορίσω τι δηλώσει και από το Συμβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ερώτησή μου που απευθύνεται και στου δύο είναι η εξή. Πότε θα ξεπεράσουμε αυτά τα πολύ ωραία λόγια, τα οποία με βρίσκουν σύμφωνοι. Πότε θα περάσουμε στην πράξη. Ε, τα ίδια λόγια τα έχουμε ακούσει πολλέ φορέ. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το Ισραήλ θα κάνει το Α, θα γίνει το Β, μάλιστα. Πώ θα καταφέρουμε κάτι τέτοιο στην πράξη. Γιατί το Ισραήλ μέχρι στιγμή μα αγνοεί. Άρα η ερώτησή μου είναι, από πρακτική άποψη, τι μπορείτε να κάνετε έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε πραγματική πρόοδο. Γιατί κατά την άποψή μου αυτό συμπεριλαμβάνει θέματα όπω για παράδειγμα η αναστολή τη Συμφωνία Σύνδεση Ευρωπαϊκή Ένωση Ισραήλ κτλ. Όσον αφορά την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Χαιρετίζω ιδιαίτερα τι πρωτοβουλίε τη Ιουδική Προεδρία και την διάβγεια όσον αφορά το ρόλο τη ε, Ιερουσαλήμ ε, ε, σαν κοινή πρωτεύουσα. Πάγωμα των επικισμών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Μάλιστα. Επίση, συμφωνώ με την έκθεση τη αντιπροσωπεία για την κατάσταση στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Και εδώ η έκθεση χαρακτηρίζεται από τη διάβγεια και το όραμα που συχνά λείπει από τέτοιε εκθέσει. Η πολιτική παράνομη προσάρτηση εκ μέρου του Ισραήλ, εσκεμμένα έχει ο στόχο να εξασθενήσει την κοινότητα των Παλαιστινίων στην πόλη. Η αρχηγοί τη αποστολή καλούν το Συμβούλιο να εγκρίνει μία σειρά από συστάσεις ως αποτέλεσμα της έκθεσης αυτής. Απαιτείται λοιπόν επίγουσα δράση από το Συμβούλιο ακριβώς για να κάνει αυτά τα οποία αναφέρονται και στην έκθεση. Εάν λοιπόν είναι σαφή η δέσμευση για την λύση των δύο κρατών, τότε θα πρέπει να, γίνει, ε, να, καταβληθεί κάθε προσπάθεια ε, για να επιτευχθούν όλα αυτά τα οποία αναφέρονται και στην έκθεση, όπου αναφέρονται και πρακτικοί τρόποι για να γίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε κυρία Λούκα και τώρα εκ μέρου των μεταρρυθμιστών και συντηρητικών για 1,5 λεπτό το λόγο έχει ο κύριο Βαντάλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φοβούνται βεβαίω ε, πάρα πολύ για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή και χάνεται η ελπίδα και νομίζουμε ότι δεν θα έρθει ποτέ η ειρήνη. Και όμως έχει σημασία όλες οι πλευρές να συνεχίσουν να εργάζονται για την ειρήνη και το πρόβλημα βεβαίως είναι θέλουν όλες οι πλευρές να εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση. Το Ισραήλ στο παρελθόν είχε κάνει το βήμα αυτό, δηλαδή γη, έναντι ειρήνης και μιλάμε εδώ πέρα για τη λωρίδα της Γάζας. Βεβαίως δεν οδηγηθήκαμε στην ειρήνη, εξακολουθήσαμε να έχουμε εχθροπραξίες και εισέβαλε τελικά το Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Τώρα ανακοίνωσε το Ισραήλ που θα σταματήσει την επέκταση των οικισμών στη δυτική όχθη του Ιορδάνη. Αυτό ως ε, κίνηση χειρονομία καλής θέλησης για τις ε, συνομιλίες που θα ακολουθήσουν. Βλέπουμε όμως πως υπάρχει μόνο κίνηση από την Ισραηλινή κυβέρνηση και δεν υπάρχει κάποια απάντηση από την Παλαιστινιακή πλευρά. Δεν υπάρχει μία ανάλογη χειρονομία. Είναι πραγματικά βούληση των Παλαιστινίων να έρθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η Χαμάς φαίνεται πως την απασχολεί μόνο ο αγώνας εναντίον της ε, Φατάχ. Ο Δε Χαμπά... Ε, Αμπάς αποδείχτηκε πως είναι ένας πρόεδρος χωρίς καμία εξουσία. Πρέπει λοιπόν και οι Παλαιστίνοι να στείλουν σαφές μήνυμα που θέλουν ειρήνη. Ευχαριστώ κύριε Βαντάλεν και το έλεγε εκ μέρου ε, τη Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά ε, για 1,5 λεπτό έχει το λόγο ο κύριο Ρετεφιλίδη. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Ήπατε, εκπρόσωπε, καλωσορίζουμε την απόφαση της 8ης Δεκεμβρίου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή επαναβεβαιώνει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δημιουργία δύο κρατών με βάση τα σύνορα του 1967 παρόλα αυτά με βάση την εμπειρία από την πρόσφατη επίσκεψή μας στην περιοχή η κατάσταση επί του εδάφους καθιστά τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους σχεδόν αδύνατη. αναφέρομαι συγκεκριμένα στην ανέγερση του τείχους στην κατεδάφιση παλαιστινιακών σπιτιών αλλά κυρίως στη δημιουργία οικισμών στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής όχθης και ιδιαίτερα στον περίγυρο της ανατολικής ιερουσαλήμ σε αυτούς τους οικισμούς ζουν σήμερα περί τους 500.000 έπικους. Ειδικότερα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ γίνεται προσπάθεια δημιουργίας κλειού με την ανέγερση οικισμών περιμετρικά της πόλης έτσι ώστε να αναγκαστούν οι Παλαιστίνοι να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους. Είναι πλέον φανερό, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση χρησιμοποιεί τις συνομιλίες για να κερδίσει χρόνο αργά αλλά σταθερά επιδιώκει την επιβολή της κυριαρχίας της επί ολόκληρου του παλαιστινιακού εδάφους. η ευρωπαϊκή ένωση θα πρέπει πέρα από την προσήλωση στη λύση δύο κρατών να αναλάβει συγκεκριμένα μέτρα έναντι του ισραήλ. η συνεχιζόμενη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί ικανή συνθήκη για να οθήσει την ευρωπαϊκή ένωση στην επιβολή κυρώσεων με βάση το άρθρο δύο της συνθήκης διότι εάν αφενό επιλέγει τη στήριξη στην επίτευξη ειρήνη αλλά αφετέρου συνεχίζει την αναβάθμιση των οικονομικών σχέσεων με το ισραήλ χωρί κανένα περιορισμό το μόνο που επιτυγχάνει είναι την εξυπηρέτηση τη πολιτική του ισραήλ που συνίσταται στον εξαναγκασμό των παλαιστινίων να εγκαταλείψουν τη γη του και την επέκταση τη ισραηλινής κυριαρχία επί ολόκληρη τη παλαιστίνη. Ευχαριστούμε κύριε Τριανταφυλλίδη. Εξ Ομάδα Ελευθερία και Δημοκρατία για δύο λεπτά το λόγο έχει ο κύριο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τρελάθηκαν στην Ευρώπη. Αυτό το ρητορικό ερώτημα μου το έθεσε ένας ε, Αμερικανός ε, συνάδελφος ε, τους μήνες που πέρασαν που θέλουν να γίνει η Ανατολική πρωτεύουσα η Ανατολική Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα του Παλαιστινιακού κράτους ε, κυκλοφορούσε ήδη τότε το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου και εγώ ως πρόεδρος αντιπροσωπείας ε, με τις ήπα ε, και του Διατλαντικού Διαλόγου είπα πως θα περιμένουμε να δούμε το τελικό ψήφισμα και θα λυπηθούν πάρα πολύ οι συνάδελφοί μου στο Κογκρέσο και εγώ θα ήθελα να αποστασιοποιηθώ από αυτό. Η δήλωση του Συμβουλίου νομίζω αποτελεί ισχυρό χτύπημα και διπλωματικό βήμα προς τα πίσω όσον αφορά την ειρηνευτική διαδικασία. Και εδώ πέρα πραγματικά πλήττεται το Ισραήλ από την Σουηδική Προεδρία. Υπάρχουν εδώ πέρα νομίζω ουσιαστικές επιφυλάξεις όσον αφορά το, ε, τα συμπεράσματα αυτά του Συμβουλίου Επίσης αναφέρεται πως δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει το κουαρτέτο στις διμερείς διαπραγματεύσεις. Πρόκειται για δήλωση της 9ης Νοεμβρίου 2008. Η δε τελευταία αμερικανική αντίδραση 8, στις 8 Δεκεμβρίου υπογραμμίζει αυτή ακριβώς την αρχή και είναι ανησυχητικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Οι δε τελευταίες μου επισκέψεις στο Ισραήλ με έπεισαν για την αναγκαιότητα μιας σταθερής και σταδιακής διαδικασίας προς το να γίνει κράτος. Το η Παλαιστινιακή Αρχή. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει στην Δυτική Όχθη του Ιορδάνη, τη λεγόμενη ζώνη Γ και θα πρέπει να οικοδομηθούν πρώτα απ' όλα οι Παλαιστινιακές Αρχές θα ήθελα λοιπόν να παρακαλώ στην Κομισιόν να μην κάνει αντιπαραγωγικέ δηλώσει για την ειρηνευτική διαδικασία και ανταυτού να επενδύσει σε συγκεκριμένα έργα συνύπαρξη Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Αυτό νομίζω πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριε Βέλντερ. Για του μη γεγραμμένους τώρα το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Ντότζ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως μέλος της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας για το Ισραήλ, με ενδιαφέρον άκουσα τα σχόλια της Προεδρεύουσα του Συμβουλίου και τη δήλωση της ε, είπα της εκπροσώπου. Ωστόσο, ο προλαλής σας ε, διατύπωσε μια ανησυχία την οποία συμμερίζομαι. Το Ισραήλ είναι η μόνη δημοκρατία που λειτουργεί στην περιοχή, ενώ η τακτική των αντιπάλων είναι η τρομοκρατία. Πιστεύω ότι συμβούλιο, οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στις προβληματισμούς ως προς την ασφάλεια του Ισραήλ. Δεν άκουσα την είπατε εκπρόσωπο να αναφέρει αυτές τις ανησυχίες. Επιπλέον, Νομίζω ότι η δήλωση επιβάλλει μεγαλύτερο βάρος στους ώμους του Ισραήλ και για την ε, πρόοδο των διαπραγματεύσεων και για την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων και ιδιαίτερως του ζητήματος της Ιερουσαλήμ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Ντότ. Και τώρα ε, να δώσουμε το λόγο στους υπόλοιπους ομιλητές. Για δύο λεπτά το λόγο έχει ο κύριο Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι η συζήτηση αυτή είναι κάπω ε, ιδιαίτερη. Γιατί από τη μια έχουμε την κυρία Μάλστρομ, εξ ονόματο του Συμβουλίου, και ελπίζουμε ε, πολύ σύντομα να τη δούμε ε, στα έδρανα τη Επιτροπή. Και πάντω, κύριε Πρόεδρε, να σα πω ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ε, δεν μας οδηγούν σε αισιοδοξία. Περισσότερο σε ανησυχία θα έλεγα, λόγω της έλλειψης προόδου όσον αφορά την ενεργητική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Ε, ε, αναφέρεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στα συμπεράσματα της συνδιάσκεψης της Μαδρίτης και στον Αττικό Χάρτη. Τίποτα το καινούριο λοιπόν. Και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι ακούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συμβάλλει για την επίλυση των προβλημάτων τα οποία ακούσαμε και εδώ, όπως τα παρουσίασαν οι δύο μιλητές. Το πρόβλημα της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, το πρόβλημα του ύδατος, το πρόβλημα της ασφάλειας, το πρόβλημα στα σύνορα. Αλλά, πρόεδρε, εδώ υπάρχει μια σειρά καινούριων προβλημάτων και εδώ θα ήθελα ε, να το τοποθετηθούν οι ομιλητριές μας. Πρώτα απ' όλα για το θέμα του μορατόριου των 8 μηνών. Ε, για το θέμα των επικισμών και την απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης. Όλα αυτά συνδέονται και με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ. Ρωτώ επίσης, ε, τι ε, πιστεύετε σε σχέση με τις δηλώσεις χτες στη Γάζα του εκπροσώπου της Χαμάς με ευκαιρία της επαιτίου που είπε ότι δεν προτίθεται να κάνουν παραμικρή υποχώρηση έναντι του Ισραήλ και να τον αγνωρίσουν. Τι, τι πιστεύετε όσον αφορά αυτό ε, το νόμο της συνέχειας και για αυτό το δημοψήφισμα για ε, τα κατεχόμενα. Και τέλος, ε, τι άποψη έχετε όσον αφορά την έκθεση Γκλάκστον και την υιοθέτησή της εκ μέρους της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Όλα αυτά είναι στοιχεία που ευνοούν την ενευτική διαδικασία ή αντίθετα όπως υποστηρίζει το Ισραήλ πρόκειται για ένα στοιχείο που δυσχεραίνει και παρεμποδίζει την ενευτική διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σαλαφράγκα και τώρα το λόγο έχει για δύο λεπτά ο κύριος Ντερόσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν δύο συγκεκριμένες δεσμεύσεις που θέλω να καλωσορίσω στη δήλωσή του Συμβουλίου που νομίζω έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μια νέα δυναμική η υποστήριξη του διετούς προγράμματος ε, της Παλαιστινιακής Αρχής για την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους και του τερματισμού της ε, Ισραηλινής κατοχής και την διαθεσιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναγνωρίσει ένα τέτοιο κράτος. Πέρσι ήμουν υπέρ της, ε, ήμουν επικεφαλής της αποστολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Παλαιστινιακές περιοχές και είδα η διεισόμαση και φέτος ε, το σύστημα Apartheid που επιβάλλεται εις βάρος των Παλαιστινίων και τους καταστρέφουν τα σπίτια, την πρόσβαση σε νερό, τη και τα λοιπά. Παρά την άδεια που είχαμε βεβαίως ως αντιπροσωπεία να πάμε στην Γάζα, αυτή ανακλήθηκε εντός ορών. Ε, δεν είναι αυτές πράξεις ενός ε, σοβαρού κράτους και οπωσδήποτε είναι παρέμβαση στο δικαίωμα του Κοινοβουλίου μας να έχουμε σχέσεις με τους δημοκρατικά εκλεγμένους Παλαιστινίους ομολόγους μας. Είδαμε την απελπισία των ανθρώπων που επισκεφθήκαμε στην Χευρώνα και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και στη Ραμάλα και όπου υπάρχει απελπισία υπάρχει βία. Μπορούμε τώρα να σημειώσουμε πρόοδο ή μπορούμε να αφήσουμε την κατάσταση να ξανακυλήσει σε χειρότερη βία που θα οθήσει και τους μετριοπαθείς Παλαιστινίους πολιτικούς να χάσουν την εξουσία. Οπότε απευθύνω έκκληση και στο Συμβουλίο και στη Βαρόνια Άστον, στην οποία έχουμε κάθε επιτυχία, να ξαναξεκινήσουν την εμπλοκή της Ένωσης στη διαδικασία αυτή και να μην τα περιμένω όλα από το κουαρτέτο. Και να θέσουν ένα χρονοδιάγραμμα που θα συμπίπτει με το διετές χρονοδιάγραμμα της Παλαιστινιακής Αρχής για την εφαρμογή των αρχών που τόσο γενναία νομίζω επαναλάβουμε την τελευταία εβδομάδα. Πρέπει να υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την πρόσβαση στις αγορές μας ως κίνητρο για το Ισραήλ. Δεν μιλάω για κυρώσει, απλά η πρόσβαση στη δική μας αγορά πρέπει να αποτελέσει κίνητρο ώστε το Ισραήλ να σέβεται τις διεθνείς του υποχρεώσεις. Και τέλος πρέπει να πείσουμε τη ΣΥΠΑ επιγόντως να επανέλθουν στη διαδικασία, στη βάση που αναφέραμε στην προηγούμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό το λόγο έχει ο κύριο Ντέβης. Πρόεδρε, η έκθεση του επικεφαλής της Αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιερουσαλήμ είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Πρώτον, η έκθεση λέει ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ανατολική Ιερουσαλήμ είναι εθνοκάθαρση. Ε, δια της βίας οι Παλαιστίνοι εκδιώκονται από τα σπίτια τους και ό,τι συνέβη για την ειρήνη καταστρέφεται. Τι πρέπει να κάνουμε. Ευπρόσδεκτες οι προτάσεις του Συμβουλίου. Ε, ε, βεβαίως η Ισραηλινή κυβέρνηση αμέσως τις απέρριψε. Τίποτα καινούριο. Και ε, βέβαια ποτέ δεν υποστηρίζουμε τα λόγια μας με πράξεις. Για ποιο λόγο. Εμείς πληρώνουμε όμως το λογαριασμό για την ε, για την, ε, για την κατοχή. Ε, οι δικοί μας φορολογούμενοι το πληρώνουν. Αν λοιπόν διακόψουμε, αναστείλουμε τη συμφωνία σύνδεσης θα, θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό θα πρέπει να σκεφτούν οι αρμόδιοι υπουργοί. Υπάρχουν τα λόγια που είναι όμως η πολιτική. Έχουμε την πολιτική, βρίσκεται στα συμπεράσματα, αλλά που είναι η δράση το Ισραήλ δεν θα κινηθεί παρά μόνο αν το σπρώξουμε. Ευχαριστούμε κύριε Ντέιβις. Τώρα το λόγο έχει για 1,5 λεπτό η κυρία Μπράτνερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλωσορίζω και την κυρία Άστον σήμερα εδώ πέρα με τη νέα της ιδιότητα. Ευχαριστώ την Προεδρία για το ψήφισμα και για την αναγνώριση του ότι χωρίς ε, τη λύση του προβλήματος των, ε, οικισμών, των επικισμών δεν θα επιτευχθεί η μακροπρόθεσμη λύση του προβλήματος. Η έκθεση του επικεφαλής αποστολής αναφέρθηκε πολλές φορές και εμείς τη βρίσκουμε θετική και έχω δύο ερωτήματα. Πρώτον, ποια είναι η τωρινή κατάσταση αυτής της έκθεσης, πού θα δημοσιευτεί. Δεύτερον, τι θα κάνει η Κομισιόν και το Συμβούλιο για να ακολουθήσει τις συστάσεις που περιέχονται εκεί πέρα. Και θα αναφέρω τρεις συγκεκριμένες συστάσεις. Η πρώτη είναι να προλάβουμε και να αποθαρρύνουμε οικονομικές συναλλαγές από κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποστηρίζουν τους επικισμούς στην Ανατολική Ιερουσαλήμ μέσω της ανάλογης ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Δεύτερον, να διασφαλίσουμε πω προϊόντα τα οποία κατασκευάζονται σε οικισμού στην Ανατολική Ιερουσαλήμ δεν εξάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω τη Συμφωνία Σύνδεση Και τρίτον, να δοθεί κάποια κατεύθυνση όσον αφορά τι ετικέτε που μπαίνουν για την προέλευση των προϊόντων. Τρει πολύ συγκεκριμένε προτάσει που γίνονται σε αυτή την έκθεση. Ποια είναι τα, τα επόμενα σα βήματα για να εφαρμοστούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μπράτνερ. Τώρα το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Λε Ιαρίκ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστώ και με ικανοποιούν τα λόγια σας. Η Ευρώπη διαθέτει δύο έγγραφα πολύ σημαντικά υπέρ νέων πρωτοβουλειών ειρήνευσης. Πρώτον, το, η θαραλέα έκθεση της Σουηδικής Προεδρίας, όπως αναφέρατε κυρία Μάλμστρομ, που ζητά να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση δύο ε, κρατών με βάση τη Συμφωνία του 67 και με την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως ε, πρωτεύουσα. Δεύτερον, ε, την έκθεση που δείχνει πώς οι Ισραηλοί προχωρούν στην κατεδάφεση των κατοικιών των Παλαιστινίων και προχωρούν σε ε, επικισμούς για να ε, κόψουν στη μέση την δυτική Όκτη. Συνεπώ, αν δεν υπάρχουν συγκεκριμένα έργα από πλευρά μα, δεν θα σταματήσει αυτή η διαδικασία. Πρέπει να δράσουμε. Πρέπει να αναστείλουμε τη Συμφωνία συνδεσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ισραήλ, εφόσον το Ισραήλ δεν σέβεται το διεθνέ δίκαιο. Χρειάζονται λοιπόν έργα κατά του επικισμού, κατά του αποκλεισμού της Γάζας, ε, ε, κατά, υπέρ της κατεδάφισης του ε, τείχους. Χρειάζονται μέτρα. Και να προσθέσω και κάτι άλλο. Μιλήσαμε για την απελευθέρωση του στρατιώτη Σαΐκ. Συμφωνώ. Αλλά ταυτόχρονα το κοινοβούλιο μας θα πρέπει να ζητήσει την απελευθέρωση και ενός άλλου Ευρωπαίου πολίτη, Γάλλο-Παλαιστίνιου, του νέου Σάλα Αμουή. Ε, ε, πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε και την απελευθέρωση του Σάλα Αμουή. Ευχαριστούμε. Τώρα το λόγο έχει για δύο λεπτά ο κύριος Μπουσούτιλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να αρχίσω επενώντας το Συμβούλιο για τα συμπεράσματα, τα θαραλέα αυτά συμπεράσματα, ε, στα οποία κατέληξε την περασμένη εβδομάδα. Νομίζω ότι ποτέ δεν είχαμε τόσο διαυγή ξεκάθαρα ε, και αποφασιστικά συμπεράσματα για ένα τόσο λεπτό θέμα εκ μέρους του Συμβουλίου. Γι' αυτό θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου ε, προ το Συμβούλιο. Θέλω να πω ότι τώρα θα πρέπει να κινηθούμε προ συγκεκριμένη δράση. Γιατί η κατάσταση στην Ιερουσαλήμ ε, πραγματικά ε, επιδεινώνεται κάθε μέρα και δεν μπορούμε να αφήσουμε να εξελίσσονται έτσι τα πράγματα. πρέπει να πούμε ότι παραβιάζεται η διεθνής νομοθεσία και ε, ε, ε, αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να είναι θύματα πάρα πολλοί άνθρωποι, να εκδιώχνονται από τα σπίτια τους τα οποία καταδαφίζονται. Δεν μπορούμε λοιπόν να ανεχθούμε πλέον αυτή την κατάσταση και να είμαστε σιωπηλοί μάρτυρες απέναντι σε τέτοια αδικία. Γιατί αν εξακολουθήσουμε να παραμείνουμε σιωπηλοί, να παραμένουμε σιωπηλοί, τότε το μήνυμα που θα εκπέμψουμε είναι ότι ε, οι βασικές αξίες ε, ε, που εμείς υποστηρίζουμε για την, για την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων δεν σημαίνουν τίποτα. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να επιτρέψουμε αυτή την κατάσταση. Αν κάτι τέτοιο συνέβαινε στη χώρα μας, τι θα γινόταν. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε και να βοηθήσουμε για την επίλυση της κατάστασης, δημιουργώντας το κατάλληλο κλίμα, το οποίο θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη και στις δύο πλευρές για την επίτευξη ε, και τη δημιουργία δύο βιώσιμων κρατών και για την εξασφάλιση της ειρήνης. Και τέλος, να αναφερθώ στο ρόλο της Ιορδανίας. Ε, που είναι πολύ σημαντικό Τέλο, απευθύνομαι προς τη Βαρόνη. Ε, Βαρόνη, έχετε τώρα ένα νέο ρόλο. Πολύ σημαντικό με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και έχουμε και εμείς την ευκαιρία για πρώτη φορά να ε, ε, συμβάλλουμε προς την επίτευξη μιας μακροχρόνιας και βιώσιμης λύσης προς τη Μέση Ανατολή. Σας παρακαλώ να μην χάσουμε την ευκαιρία αυτή. Για 1,5 λεπτό τώρα το λόγο έχει ο κύριος Κροτσέτα. Ε, ε, ε, κοιτάξτε, Πρόεδρε, ήμασταν στη Ραμάλα όταν έφτασε η πληροφορία ότι η Ευρώπη πήρε μια νέα απόφαση για την ενευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Είδαμε τα χαμόγελα και τι ελπίδε στου Παλαιστίνιου. Οι μέρε αυτέ ήταν γεμάτε ένταση και πραγματικά αισθανθήκαμε τρομερή αγανάκτηση όταν είδαμε τα παιδιά, την κατάσταση των παιδιών σε αυτού του δρόμου φαντάσματα που δεν μπορούσε να, τη που δεν μπορούσε να περάσει κανένα άνθρωπο. Είδαμε μια γυναίκα 80 χρονών να τη διώχουν από το σπίτι τη και να κοιμάται σε μια σκηνή ε, στον κήπο αυτού που, ε, στο, σε αυτό που κάποτε ήταν ο κήπο τη και να ε, κοιμάται μέσα στο κρύο. Με κονδύλια λοιπόν, με ευρωπαϊκά κονδύλια είχε, δημιουργηθεί, είχε χτιστεί ένα εργοστάσιο το οποίο το κατέστρεψαν οι Παλαιστίνοι, οι, οι, οι Ισραηλοί, συγγνώμη. Το Ισραήλ έχει δικαίωμα σε ένα κράτο, αλλά το ίδιο δικαίωμα έχουν και οι Παλαιστίνοι. Η απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης αποτελεί σημαντικό βήμα προς τα, του Ευρωπαϊκού του Συμβουλίου αποτελεί σημαντικό βήμα, αλλά θα πρέπει να ε, γίνει κι άλλο ένα βήμα. Γιατί εδώ μιλάμε για την κορυφή του παγόβουνου μιας ευρύτερης σύγκρουσης. Τις ε, τελευταίες ημέρες ε, πρόσφατα μας παρεμπόδισαν οι Ισραηλινές αρχές να επισκεφθούμε τη λωρίδα της Γάζας. Ε, παρεμπόδισαν την αποστολή του Κοινοβουλίου. Και νομίζω ότι η Βαρόνι Άστον, ε, είπα εκπρόσωπος, θα πρέπει να παρέμβει και να εκφράσει τη διαμαρτυρία της Ευρωπαϊκής ε, της Δημοκρατικής Ευρώπης. Ευχαριστώ και τον πρόεδρο της Αντιπροσωπείας, τον κύριο Ντερόσα και τα άλλα μέλη της Αντιπροσωπείας, διότι ε, τις ημέρες εκείνες που βρεθήκαμε στην Παλαιστίνη ε, μπορέσαμε να δούμε την κατάσταση επι, επιτόπου. Να, ε, και οι Παλαιστίνοι είδαν το πρόσωπο μιας Ευρώπης που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των πολιτών και που θέλει να συμβάλλει περισσότερο για την ε, επίτευξη λύσης. Ευχαριστούμε τώρα ε, και δίνουμε το λόγο για ένα λεπτό στον κύριο Τακούλη. Πρόεδρε, είπατε εκπρόσωπε. Είμαι βέβαιος ότι είπατε εκπρόσωπος ε, διαρωτάτε τι κάνουμε εμείς ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι ιστορία διαβάζουμε. Δεν ξέρουμε ότι το, Ισραήλ, το κράτος του Ισραήλ ιδρύθηκε το 1947. Η σουηδική στάση είναι κάπως περίεργη. Πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη και να τηρούμε τις αξίες μας. Έχουμε δημοκρατία, ε, ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερία. Το Ισραήλ είναι το μόνο δημοκρατικό κράτος ε, στη Μέση Ανατολή δεν πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε άλλε χώρε οι οποίε ε, δεν είναι δημοκρατικέ και δεν συμμερίζονται τι δικέ μα αξίε. Η ιδέα του διαχωρισμού τη Ιερουσαλήμ ω πρωτεύουσα ε, δύο κρατών είναι κάτι το ακατανόητο. Δεν είναι λύση αυτή. Θα πρέπει να προσέξουμε ώστε το Ισραήλ να διατηρήσει τη δημοκρατία του, να έχει το δικαίωμα στη δική του πρωτεύουσα. Και από την άλλη η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εμπλακεί στην ενευτική διαδικασία. Είναι υποχρεωτικό, αλλά ως διπλωμάτης, ως, ως διπλωμάτης όχι ως κριτής, ως δικαστής ως, ως γιατρός και όχι ως δικαστής. Πρόεδρε, είναι πραγματικά δυσάρεστο που δεν έχει απελευθερωθεί ο Ισραηλινός στρατιώτης. Αυτό μας δείχνει το πώς η Χαμάς βλέπει τις δικές μας αξίες. Πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθούμε και να απορρίψουμε αυτές τις άχρηστες ιδέες που περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Το Ισραήλ είναι μια δημοκρατία, συμμερίζεται τις αξίες μας, μοιράζεται τις αξίες μας και εμείς πρέπει να σεβαστούμε το δικαίωμα των ανθρώπων να ζήσουν εν ειρήνη εκεί. Η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί όταν τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Χαμάς και άλλες θα σταματήσουν τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τους τρομοκράτες και να δημιουργήσουμε τη δυνατότητα ύπαρξης στον Ισραηλινό λαό. Ευχαριστώ κύριε Τακούλα. Για ένα λεπτό έχει το λόγο κυρία Μπρέπολ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο επικεφαλής αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιερουσαλήμ και στη Ραμάλα ή επικεφαλής ξεκαθάρισαν στην έκθεση της 23 Νοεμβρίου πως ε, προσαρτά παράνομα το Ισραήλ την Ανατολική Ιερουσαλήμ που πρέπει να κάνει το ίδιο και με την υπόλοιπη δυτική όχθη. Γιατί δεν βγάζει τα σωστά συμπεράσματα εδώ πέρα το Συμβούλιο. Γιατί μια τόσο σημαντική έκθεση δεν ε, ακολουθεί μετά τα συμπεράσματα και τις συστάσεις που αναφέρονται. Δηλαδή οι εξελίξεις αυτές θα καταλήξουν να είναι μετά μη ε, Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος. Πλέον δεν έχει νόημα να κάνουμε κενές δηλώσεις πρέπει να παίξουμε έναν ενεργό και ορατό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην περιοχή ως Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό γίνεται με το να βρούμε το θάρρος πρώτα απ' όλα να πούμε τα πράγματα με το όνομά της και οπωσδήποτε όσον αφορά την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Ευχαριστώ κύριε Μπρέπελς. Για ένα λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Αγκουράκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η πολιτική της ευρωπαϊκής ένωσης είναι αυτή που μαζί με τις ηνωμένες πολιτείες και το νατο στηρίζουν την ισραηλινή κυβέρνηση στην εγκληματική πολιτική της γενοκτονίας του παλαιστινιακού λαού. αυτό είναι το συμπέρασμα βουλευτών που συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου που οι αρχές του ισραήλ απαγόρευσαν την είσοδο στην κατεχόμενη λωρίδα της γάζας. η πολιτική της ευρωπαϊκής ένωσης και η τελευταία απόφαση του συμβουλίου ουσιαστικά δίνουν χρόνου στις ισραηλινές κυβερνήσεις που βαραίνονται με εγκλήματα πολέμου όπως ξέρουμε από την έκθεση του οηε για τον πόλεμο στη γάζα για να συνεχίσουν το κατοχικό του σχέδιο. τα μασημένα λόγια της ευρωπαϊκής ένωσης δεν ανταποκρίνονται στο δίκαιο παγκόσμιο αίτημα για βιώσιμο και ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος στα εδάφη του 1967 με πρωτεύουσα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λαμβάνει κανένα πρακτικό μέτρο σε αυτή την κατεύθυνση. Αντίθετα, αναβαθμίζει τι σχέσει με το Ισραήλ, που συνεχίζουν τους επικισμούς ιδίως στην Ανατολική Ιερουσαλήμ την κατασκευή διαχωριστικού τείχους του έσχους τον ε, εγκληματικό αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας. Αποκρούμε τα εμπεριλαστικά σχέδια για τη Μέση Ανατολή και συμπαριστοκόμαστε ολόπλευρα στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού και των όλων λαών της περιοχής. Ευχαριστούμε κύριε Αγγουράκη. και τώρα το λόγο έχει για 1,5 λεπτό η κυρία Φλασίκοβα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της ε, προηγούμενης εβδομάδας ε, είναι σαφή, ξεκάθαρα. Νομίζω πως ξέρετε πως ασχολούμαι καιρό με αυτό το ζήτημα. Δεν έχουμε επιτύχει σημαντική πρόοδο. Θα ήθελα λοιπόν να υπενθυμίσω ακόμη μία φορά πως ε, γνωρίζουμε πως ε, πρέπει να παίξουμε έναν ενεργό διαμεσολαβητικό ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία. Πρέπει να επιμείνουμε να ξεπεραστεί αυτή η καταστροφική και για τις δύο πλευρές ε, κατάσταση έτσι ώστε οι Παλαιστίνοι και το Ισραήλ ε, να εμπλακούν στην ε, διαδικασία. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε και από τους ε, Παλαιστίνιους να επανέλθουν στις διαπραγματεύσεις. Επιμένουμε πως θα πρέπει να φύγουν τα εμπόδια, δηλαδή η οικοδόμηση στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, το τείχος, όλα αυτά είναι απαράδεκτα είναι απαράδεκτο το Ισραήλ να μην μπορεί όμως να αντιδράσει και σε τρομοκρατικές ενέργειες. Θα ήθελα να υπογραμμίσω πως ε, πράγματι πρέπει να γίνει σεβαστό και το διεθνές δίκαιο. Θεωρώ λοιπόν πως εμείς οι Ευρωπαίοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολίτες είμαστε διατεθειμένοι να απλώσουμε το χέρι μας για την ειρήνη. Θα ήθελα λοιπόν να ευχηθώ επιτυχία και στην κυρία Άστον και να μας φέρει μια μέρα θετικά νέα. Ευχαριστώ, κυρία Φλάσικοβα. Η κυρία Τάιν έχει το λόγο για ένα λεπτό. Κυρία Υπουργέ, κυρία εκπρόσωπε, Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι μέλος της ε, αποστολής για τις σχέσεις με το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο δηλαδή της Παλαιστίνης. Δεν μπορέσαμε να πάμε στη Γάζα την προηγούμενη εβδομάδα, μας το απαγόρεψε το Ισραήλ, είναι ανισχυτική η κατάσταση στη Γάζα, ειδικά τώρα το χειμώνα, μόνο 10% του πληθυσμού μπορεί να συντηρηθεί και μιλάμε ε, ε, ότι πρόκειται κυρίως για λαθρεμπόριο μέσω των τούνελ η δε κατάσταση πριν από την επιχείρηση Βαρύ Μολύβη ήταν ε, αντίστροφη. 90% μπορούσε να συντηρήσει τον εαυτό του. Θα πρέπει λοιπόν να ανταποκριθεί το Ισραήλ στις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το διεθνές ε, δίκαιο. Αλλιώς να επέμπει η Διεθνή κοινότητα και κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν όμως είναι το Ισραήλ να φροντίσει να φροντίζει για το 90% του πληθυσμού, θα πρέπει να δούμε και εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση πού πάνε τα λεφτά τα δικά μα των Ευρωπαίων φορολογουμένων, εάν ξοδεύονται σωστά. Ευχαριστούμε. Και τώρα το λόγο για ένα λεπτό έχει η κυρία Φλότ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία μάστρομ και την Σουηδική Προεδρία για τα συμπεράσματα τα οποία επαναλαμβάνουν ακριβώς αυτό που αναμένουμε, δηλαδή την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ειρήνη στην περιοχή επί τη βάση της διεθνούς, της διεθνούς και αυτό είναι θεμελιώδη σημασίας. Ωστόσο, ένα χρόνο μετά τη στρατιωτική εισβολή στη Γάζα δεν υπάρχει αναφορά σε αυτά τα συμπεράσματα και συνέχεια της έκθεσης Goldstone. Πού βρισκόμαστε σε σχέση με την έκθεση Goldstone πάνω στο οποίο δεσμεύθηκε το Συμβούλιο όσον αφορά την εσωτερική έρευνα ή τις εσωτερικές έρευνες των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών. Δεύτερον, ε, χαίρομαι που αναφέρεται η Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Παλαιστινιακού κράτους ή πρωτεύουσα των δύο κρατών. Ωστόσο, ε, από τα συμπεράσματα αυτά δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις ως προς ε, το πώς θα ρυθμιστεί αυτό. Ζητώ λοιπόν από την Κομισιόν και το Συμβούλιο να διευκρινίσουν τις συγκεκριμένες ενέργειες ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην αναγνωρίσει ή να μην ονειμοποιήσει την ε, ε, τις διαδικασίες που ακολουθεί το Ισραήλ και τα Ανατολική Ιερουσαλήμ και στα οικονομικά αλλά και τη μαζική μεταφορά ε, Παλαιστινίων από την περιοχή. Ευχαριστώ για να λεπτό το λόγο ο κύριος Χόβιτ. Χαιρετίζω, καλωσορίζω την ύπατη εκπρόσωπο στην ε, ολομέλεια αλλά επίσης και την ισχυρή θέση του Συμβουλίου. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον κύριο Μπίλτ εξ της Προεδρίας για το γεγονός για την αξιοπιστία και την ε, αποτελεσματικότητα της έκθεσης ε, και όπως ακριβώς είπε ο ε, πρεσβευτής στον ΟΗΕ η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ζητά να υπάρξουν αξιόπιστες έρευνες σχετικά με τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέλος θα ήθελα να ρωτήσω την Προεδρία και την είπα ότι εκπρόσωπο γνωρίζουν την ε, οδηγία της Βρετανικής κυβέρνησης για ειδική σήμανση των, σε τρόφιμα που προέρχονται από τις Παλαιστινιακές τα παλαιστινιακά κατεχόμενα εδάφη και τι σχέδια υπάρχουν ώστε αυτό να επεκταθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, εμείς ως Ευρωπαίοι ε, πληρώνουμε το κόστος και ως καταναλωτές δεν πρέπει να επιδοτούμε. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό κύριε Στρεμός έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι η πρόσφατη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με βάση ε, την πρόταση της Σουηδικής Προεδρίας, ε, υπό την καθήκηση της Σουηδικής Προεδρίας μάλλον, για την Ιερουσαλήμ ως κοινή πρωτεύουσα, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά την προσπάθειά μας, τη διαμεσολαβητική προσπάθεια μπορεί να είναι αντιπαραγωγική σε σχέση με το βασικό στόχο, την επίτευξη της ειρήνης σε αυτή ε, την ε, δοκιμαζόμενη περιοχή. Νομίζω ότι αντί να ακολουθούμε αυτή αυτή την μονομερή και απρόσμενη οδό ανακοίνωση μιας πρότασης, θα ήταν καλύτερο και πιο χρήσιμο η Ευρωπαϊκή Ένωση να συγκεντρώσει όλες τις προσπάθειες ε, στην ενθάρρυνση ε, προς την κατεύθυνση της δημιουργία μιας πραγματικής και της εγκαθίδρυσης μιας πραγματικής δημοκρατίας ε, στην, στην Παλαιστίνη. Με αυτόν τον τρόπο, όπως για παράδειγμα υποστήριξη τη μη βίαιη αντιπολίτευση έτσι ώστε να υπάρχει ένα αξιόπιστο πιστό ε, συνομιλητή. Και όπω είπε και η κυρία Μάλστρομ σήμερα, ε, το θέμα τη Ιερουσαλήμ ε, θα είναι από τα αντικείμενο διμερού διαπραγμάτευση ανάμεσα στι δύο πλευρέ. Αντί λοιπόν να έχουμε μία λύση δύο κράτη για δύο λαούς, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για δύο δημοκρατίε, για δύο λαού. Η δημοκρατία, αγαπητοί συνάδελφοι, αποτελεί απαραίτητη προπόθεση για την επίτευξη τη ειρήνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Τρεμόσα. Και τώρα περνάμε ε, στι παρεμβάσει Catch the Eye. Ε, λοιπόν, προχωράμε στη διαδικασία Κάσης διάει. Ο κύριος ε, Γκέλλερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι για το ότι η Βαρόνια στον κάθισε στην πλευρά της Κομισιόν. Ελπίζω και στο μέλλον να συμβαίνει αυτό. Κατά τα λοιπά, έχω μία ερώτηση προς την Προεδρία του Συμβουλίου. Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών λείπει μία αναφορά στο κουαρτέτο. Δεν συμφωνείτε με το ρόλο του κουαρτέτου. Ποιος είναι ο λόγος, αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Δεύτερον, το ίδιο ισχύει και για την Χαμάς και για αυτή την δυστυχώς πολιτικά σημαντική ομάδα δεν υπάρχει κάποια αναφορά. Ποιος είναι ο λόγος. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, ε, θα προσπαθήσω ε, να μην ε, μιλήσω και μακρηγορήσω. Πάντως σας πω το εξή. Η Σουηδική Προεδρία μας είχε συνηθίσει σε πολύ περισσότερα από αυτά και ζητώ συγγνώμη κυρία Μάλστρομ τα οποία αποφασίστηκαν όσον αφορά την Ιερουσαλήμ. Κοιτάξτε, αυτό αποτελεί διπλωματικό σφάλμα κατά την άποψή μου, το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο. Όχι επί τη ουσία. Μην παρεξηγήσετε αυτά τα οποία αναφέρω, αλλά όσον αφορά τη δήλωση αυτή που προδικάζει το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Ε, και αυτό ε, μπορεί να το θεωρήσουν ω ε, προσβλητικό και οι δύο πλευρέ. Ε, γι' αυτό, κοιτάξτε, ε, ε, ε, ορισμένοι πήραμε τι αποστάσει μα όσον αφορά τη δήλωση αυτή. Βεβαίω, συμφωνούμε. Μια ανοιχτή πρωτεύουσα, μια κοινή πρωτεύουσα από το 2000 αυτό το κοινή πρωτεύουσα συμπεριλαμβάνεται στι παραμέτρου Κλίντον. Ε, πρόκειται για μια αρχή την οποία την, είχε, ε, την είχαν δεχθεί ε, πολλοί ηγέτε και μην ξεχνάμε και αυτά τα οποία είχαν αναφερθεί και στο παρελθόν. Βεβαίω η Αγία Πρωτεύουσα, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, πρωτεύουσα ελεύθερη, ανοιχτή. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να επιβάλλουμε το, το μοίρασμα, το χρονοδιάγραμμα, του τρόπου, τι λεπτομέρειε εφαρμογή εφαρμογή, αλλά όπω αναφέρθηκε προηγουμένω, να ενθαρρύνουμε το διάλογο έτσι ώστε οι Παλαιστίνοι και οι Ισραηλοί να καταλήξουν ένα συμπέρασμα. Σα ζητώ συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, αλλά ορισμένοι ομιλητέ διπλασίασαν το χρόνο αγόρευση. Εγώ έχω ένα λεπτό, δεν μπορεί εδώ να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν με ενδιαφέρει πόσο μίλησαν οι προηγούμενοι ομιλητέ. Εγώ σα έδωσα ένα λεπτό, ένα λεπτό θα μιλήσετε. Ζητώ συγγνώμη ε, στου υπόλοιπου γιατί σα έδωσα μισό λεπτό παραπάνω. Δεν πρόκειται να ξανασυμβεί. Θέλω επίση να πω και στου υπόλοιπου ότι έχω πέντε ονόματα μπροστά μου Δυστυχώ δεν έχουμε χρόνο. Ζητώ συγγνώμη από όσου δεν θα μπορέσουν να μιλήσουν στη διαδικασία Catch the Eye. Κυρία Λάτφορντ, για ένα λεπτό, επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου είναι πρόσδεκτα σχετικά με τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πρόθεση να διαδραματίσει ισχυρότερο ρόλο για να επαναδραστηριοποιηθεί το κουαρτέτο. Συμφωνεί το Συμβούλιο και η Κομισιόν ότι η προσέγγιση κάποιων να μποϊκοτάρουν το Ισραήλ είναι εσφαλμένος δρόμος για αυτή την εμπλοκή. Δεν μπορεί κανείς να μποϊκοτάρει και να εμπλέκεται ταυτόχρονα. Η σωστή προσέγγιση είναι αυτοί που προτείνουν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, δηλαδή περαιτέρω ανάπτυξη δημερών σχέσεων με το Ισραήλ που επιβεβαιώνονται. Όσο ε, και μπαίνει στον πειρασμό, το Συμβούλιο έχει επιρροή πολιτικά και οικονομικά, οικονομική υποστήριξη και αντιστέκεται σε αυτόν τον πειρασμό τους πειρασμούς που προέρχονται από των διαφόρων μερών ώστε να προτείνουν και Ρώσοι στη μία ή την άλλη πλευρά. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ σύνθετη και ε, θα υπονόμευε μια συνεκτική ε, συνεπή ε, στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να υπάρξει τελικά ειρηνευτική συμφωνία. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. και πρέπει να πω ότι δεν είμαι υπέρ των κυρώσεων και των απειλών, είμαι υπέρ επικοδομητικής πολιτικής και διαλόγου. Ωστόσο φοβούμε ότι πάρα πολύ συχνά, όπως λέγεται εδώ, ελέγχθη εδώ ότι το Ισραήλ είναι δημοκρατικό κράτος, αλλά ως κράτος δεν συμπεριφέρεται δημοκρατικά όσον αφορά στους Παλαιστινίους ή στο κοινό μας στόχο και σκοπό που είναι η ίδρυση δύο ασφαλών δημοκρατικών κρατών που θα ζουν το ένα δίπλα στο άλλο. Και κυρία Μάλστρομ, Ακούσατε πολλές προτάσεις εδώ για πιο αποτελεσματική και επικοδομητική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δυστυχώς το Ισραήλ ουσιαστικά βλέπει ως ε, προσχηματική απειλή και όχι σοβαρή για να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και να επιληθεί το ζήτημα. Ευχαριστώ. Not here. Mr. Not here. Ο κύριος Άτκινς για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ως μέλος της αντιπροσωπείας που πήγε στην Παλαιστίνη, την προηγούμενη εβδομάδα κατέστησε σαφές πως υπάρχουν πολλοί λογικοί άνθρωποι που θεωρούν πως η λύση των δύο κρατών είναι τελειωμένη υπόθεση. Κύριος λόγω Ισραηλινών δράσεων ε, για επέκταση του τείχου εντός της Ανατολικής Ιερουσαλήμ επεκτείνοντας έτσι το χάσμα και το τι σκοπεύουμε να κάνουμε εάν καταλήξουμε σε ένα κράτος. Δεύτερον, η Προεδρία και οι Λέδη Άστον γνωρίζουν τις απόψεις των λογικών ανθρώπων για την παροδία αυτή που λέγεται ε, κουαρτέτο τι σκοπεύουμε να κάνουμε για να είναι το αποτέλεσμα αυτής της υπόθεσης ανάλογο του κόστους γιατί αυτή τη στιγμή είναι μηδέν το αποτέλεσμα Εκτός μικροφώνου. Ε, κοιτάξτε, ε, ε, τελικά η τελική δήλωση του, του Συμβουλίου είναι ίσως καλύτερη από την προηγούμενη εκδοχή που είχα δει πριν από λίγε εβδομάδε. Αλλά δεν αναφέρεται στη, σε αυτά τα οποία πρεσβεύει η Χαμάς και το τι ακριβώ γίνεται στη Γάζα. Επίση, γιατί ο υπουργό Εξωτερικών, ο κ. Μπίλ, δεν επισκέφτηκε την περιοχή για να δείξει την αλληλεγγύη προ το Δημοκρατικό Ισραήλ και του Μητροπαθείς Παλαιστινίου. Κάτι άλλο. Γιατί η Τη της Ανατολικής ε, ε, Ιερουσαλήμ αναφέρεται μόνο αυτό το θέμα. Πρέπει η δράση μας να χαρακτηρίζεται από ισορροπία και να προωθεί τις κοινέ δημοκρατικές αξίες και να ενισχύσει ε, τη συμμετοχή του Ισραήλ στα προγράμματα του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνώ με την Βαρόν Λάντφορντ. Πρέπει να δημιουργήσουμε κλίμα εμπιστοσύνη στη σχέση με το Ισραήλ και να δείξουμε ότι έχουμε καλή θέληση. του Συμβουλίου, κυρία Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσω και για την πολύ καλή συζήτηση. Θα ήθελα να ξεκινήσω με κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις και μετά να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Για την έκθεση Goldstone είναι πολύ σημαντική έκθεση, σοβαρή έκθεση και σημαντικό είναι να δούμε συγκεκριμένα και λεπτομερώς τα συμπεράσματα. Καλούνται και οι Παλαιστίνοι και οι Ισραηλινοί να ερευνήσουν λεπτομερώς ε, τα πράγματα. Για το κουαρτέτο τώρα. Υπάρχει αναφορά στο κουαρτέτο και στην ε, ανάγκη δραστηριοποίησης του όσον αφορά δε, την ε, Χαμάς, οι συνεχιζόμενες συζητήσεις του Συμβουλίου με τους κυρίους ε, Φαγιάντα ε, και Αμπάς ε, είναι συνεχές και είναι σαφής, σαφές το ότι δεν υπάρχει πλήρης ικανοποίηση τώρα. Σαφώς έχουν υπάρξει κάποιες αποχρώσεις όσον αφορά την στάση μας, αλλά υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση όσον αφορά τη στήριξη της ειρηνευτικής ε, διαδικασίας. Ε, ξέρετε πως ε, πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, αλλά δεν ξέρουμε αν θα έρθει επιγής ειρήνη, τουλάχιστον σε εκείνο το κομμάτι της γης. Ξεκινήσαμε τη Σουηδική Προεδρία με τις δραστηριότητες του Πρόεδρου Ομπάμα όσον αφορά τις διαπραγματεύσει Παλαιστινίων Ισραηλινών και πρέπει να συνεργαστούμε στενά με τι ΣΥΠΑ. Δεν έχει συμβεί ε, αυτό ακόμα. Βεβαίω σε αυτό το ζήτημα πρέπει να είμαστε επίμονοι και υπομονετικοί. Πρέπει να παραμείνει σταθερή η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα μηνύματα τα οποία στέλνει για την Ανατολική Ιερουσαλήμ, για του επικισμού, ε, για τα συνοριακά φυλάκια κτλ. Χαίρομαι για τη στήριξη που υπάρχει εντός του Κοινοβουλίου για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ε, και έγινε κατανοητή νομίζω και θα αποτελέσει τη βάση για το μελλοντικό έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Τώρα για τις ε, αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην περιοχή. Προσπαθήσαμε να υποστηρίξουμε τα μέτρα ειρηνευσική ασφάλεια στην περιοχή για να υπάρξει μια προετοιμασία ανεξαρτητοποίησης του Παλαιστινιακού κράτους. Υποστηρίζουμε το Παλαιστινιακό σχέδιο για να τελειώσει η κατοχή και να ανακηρυχθεί ανεξάρτητο κράτος η Παλαιστίνη. Τώρα, για να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα στην κατάσταση, πρέπει να συμφωνήσουμε. Δεν είναι ανάγκη να περιέχονται τα πάντα σε μία λύση, ούτε χρειάζονται μονομερείς ε, λύσεις και τελεσμένα. Πρέπει να είναι η λύση συνολική, να περιλαμβάνουν και κάποια πράγματα για την Συρία και το Λίβανο, να υπάρξει μια γενικότερη αντιμετώπιση της Ισραηλινο-Αραβικής ε, σύγκρουσης, οπότε υπάρχει αρκετά μεγάλο βαθμό ε, συμφωνίας, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και στήριξη των λοιπόν δεσμικών οργάνων και αναμένω τη συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστώ. Έχει ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι στη θέση αυτή είμαι βέβαιη ότι θα έρχεται και θα επανέρχεται το θέμα αυτό. Ε, και βεβαίως κάθε φορά που ε, ε, ενδεχομένως αν βρισκόμουν στην άλλη πλευρά της, ε, του καθίσματος θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ευχαριστώ πάντως τη Σεσίλια για την δική της παρέμβαση. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Πράγματι υπάρχει μια πεποίθηση την οποία συμμεριζόμαστε για μια λύση δύο κρατών. Και πράγματι από τους περισσότερους βουλευτές και ιδιαίτερα τον κύριο Ντερόσο και από τα μέλη που έλαβαν το λόγο υποστηρίζεται η θέση αυτή ακριβώς επειδή είδαν την φοβερή κατάσταση που επικρατεί επί τόπου. Τώρα, τα συμπεράσματα νομίζω ότι είναι απόλυτο σαφή και νομίζω ότι μου δίδουν και μια κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να προχωρήσουμε. Και είναι επίσης σαφές και εκτιμώ το έργο που έκανε η Προεδρία είναι σαφές ότι επικρατεί μια απογοήτευση στο σώμα αυτό ότι τα πράγματα δεν προχωρούν ε, και παρά το γεγονό ότι υπάρχουν διαφορετικέ απόψει, ο στόχο είναι ενιαίο. Να υπάρξει λύση. Να υπάρξει ε, συνδυασμό των διαφορών αλλά και των ομοιοτήτων ε, που υπάρχουν μεταξύ μα, ώστε να προχωρήσουμε στις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις. Δεν έχω αμφιβολία ότι θέλουμε δύο πράγματα. Πρώτον, τα πολιτικά ζητήματα Ποια είναι η σχέση μας, ποια πρέπει να είναι. Βρίσκομαι στην αρχή αυτού του ταξιδιού και η συζήτηση αυτή είναι εξαιρετικά χρήσιμη για μένα να ακούσω αυτές τις απόψεις που διατυπώθηκαν. Πρώτον, ότι πρέπει το κουαρτέτο να αποδείξει ότι αξίζει τα λεφτά του. Θα πρέπει να ξαναζωντανέψει. Και έκανα μια ε, ε, συνομιλία με τον κύριο Τόνι Μπλερ και είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να αναζωογονηθεί το έργο του κουαρτέτου. Δεύτερο, τα θέματα στην περιοχή που έθεσε και η Προεδρία, τα ευρύτερα ζητήματα, οι άλλες χώρες που πρέπει να εμπλακούν. Και το πιο σημαντικό που προέκυψε από τη σημερινή συζήτηση τι πρόκειται να κάνει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τούτο με φέρνει σε αυτό που αποκαλώ το πρακτικό πεδίο. Διάφοροι συνάδελφοι έθεσαν επιμέρους θέματα σχετικά με τη σήμανση, σχετικά με τη συμφωνία σύνδεσης, σχετικά με την έκθεση αν είναι επαρκής και αν οι συστάσεις που δεν έχουν ακόμα μελετηθεί ε, ε, ισχύουν ή όχι. Όλα αυτά τα ζητήματα. Πάντως πρέπει να επιδείξουμε την πρακτική υποστήριξη, υποστήριξη που απαιτείται. Ε, ε, εμείς υποστηρίζουμε το έργο του Πρωθυπουργού ε, Φαγιάτ. Θέλουμε πρακτικά να εμπλακούμε στο χώρο και να συνεργαστούμε ώστε η κατάσταση να βελτιωθεί για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να ζουν εκεί καθημερινά και οι οποίοι προσβλέπουν στη βοήθεια που χρειάζονται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και πρακτικό πράγμα που θέλω να κάνω. Θα περιγράψω το έργο μου ως εξής. Έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε πολιτικά και οικονομικά. Αυτό που θέλω είναι να συνδυάσω τα δύο πράγματα, να βρούμε έναν τρόπο να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο αυτό που κάνουμε, να γίνει πιο αποτελεσματικό το κουαρτέτο, Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λειτουργούν ο ένας στο πλευρό του άλλου και όλα αυτά μαζί να γίνουν ενιαία. Τελικά, οι δύο πλευρές πρέπει από κοινού να λάβουν μια απόφαση και να αναζητήσουν την ειρήνη. Όμως, ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε σημαντικό ρόλο να παίξουμε και είμαι αποφασισμένη εξ ονόματό σα και εξ ονόματο του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα διαδραματίσω αυτό το ρόλο. Ευχαριστώ. Ε, λίγη συζήτηση για αυτό το θέμα. Η ημερήσια διάδεξη προβλέπει συζήτηση για προφορικές ερωτήσεις σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα με αντίκτυπο στα δεδομικά δικαιώματα κατόπιν της θέσης σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Ε, αρχίζουμε τη συζήτηση με την κυρία Μποσκούρτ για τρία λεπτά.